Κυρίε και κύριοι, άρχονται οι ψηφοφορίες. Θα σας παρακαλούσα, θέλετε να καθίσετε. Πριν την έναρξη των ψηφοφοριών έχω ε, το θλιβερό καθήκον να σας κάνω μια πάρα πολύ δυσάρεστη ανακοίνωση. Στις 24 Νοεμβρίου 112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τρομερή πυρκαγιά στην Τάκα, την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, ε, σε μια κλώστο εφαντοργία. Δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου, τα μέτρα προστασίας και τα αντιπυρικά ήταν ακατάλληλα, τα δε υλικά έφλεκτα και όλα αυτά συνέβαλαν σε αυτή τη καταστροφή και τη συμφορά. Τώρα, όπως είναι λογικό, αυξήθηκε η λαϊκή δυσφορία απέναντι σε αυτή τη θεομηνία. Ε, χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν βγει στους δρόμους στην Τάκα και ζητούν καλύτερη προστασία. Στην κηδεία συμμετείχαν 100.000 άνθρωποι. Και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να ε, κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτή την τραγωδία. Στο Βαγκλαντές υπάρχουν πάνω από 4.000 κλωστοϊφαντουργίες και οι περισσότερες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Οι περισσότερες εξαγωγές ε, απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πολύ συχνά πρόκειται για μεγάλες εμπορικές μάρκες πάρα πολύ γνωστές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διερευνηθεί αυτή η τραγωδία, ε, οι συνθήκες εργασίας ε, που επικρατούν στη χώρα, τον Μπαγκλαντές, και επίσης φρονείω ότι χρειάζεται να αναλυθούν επιπτώσεις σε σχέση με μελλοντικές ε, εμπορικές συμφωνίες. Αντί λοιπόν να συζητηθεί αυτό το θέμα ως κατεπήγον, όπως είχε προβλεφθεί για την παρούσα εβδομάδα, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει πλήρη συζήτηση για το θέμα αυτό στη Σύνοδο του Ιανουαρίου, ε, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων ε, Συμβουλίου και Επιτροπής. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων ημών εκφράζω τα πιο ειλικρινά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ε, στους ε, εγκαυματίες και στους τραυματίες για πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Στη συνεδρίαση της 20ης Α, δεύτερη ανακοίνωση, τελείωσε η πρώτη. Στην συνεδρίαση της 22ης Νοεμβρίου 2012 η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε σύσταση σε σχέση με ε, τη λήξη της εντολής της ειδική Επιτροπής ε, για το οργανωμένο έγκλημα, τη ε, διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που Εκπνέει η εντολή αυτή κανονικά στις 31 Μαρτίου του 2013 και προτείνεται παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 184 του κανονισμού. Διαφωνεί κανεί, Αν όχι, εγκρίνεται η διεύρυνση αυτή τη εντολής και η παράταση λειτουργία τη Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ούτω λοιπόν και αποφασίζεται. Μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η εντολή τη Επιτροπή το 2013. Τελευταία ανακοίνωση. Ορίστε. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, από ευκαιρία της παράτασης των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής,